Έχω λάβει από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών μία, ένα αίτημα για να ε, διοριστεί ο κ. Τσάς στη θέση του κ. Ξασνοντεύσκη ως μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης. Διαφωνεί κανείς? Όχι και σας ευχαριστώ πολύ.